Λοιπόν, έγινε μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, το λέω για όσους έρχονται τώρα. Η συνάντηση με την νομική υπηρεσία θα γίνει στις 12 και θα ψηφίσουμε το σημείο 13. Εμείς προσαρμόσαμε τη γνωμοδότηση του ψηφίσματος. του προϋπολογισμού έχουμε μία τροπολογία Και θα ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία υπέρ. Λοιπόν, καλά που μου τα λέτε γιατί εγώ είμαι καινούργια. Λοιπόν, κατά, κανένας, αποχές, κανένας. Εγκρίνεται λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν θα ψηφίσουμε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Πολύ ωραία λοιπόν αυτό. Με την ομοφωνία. Στο επόμενο σημείο τώρα. καταπολέμηση της φτώχειας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι αυτό, το συζητήσαμε και σύντομα θα εγκριθεί και η ε, σχετική έκθεση. Είναι σαφές ότι χρειάζεται υποστήριξη στην ανάπτυξη και είναι και ο μεγαλύτερος δωρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να τεθούν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το, τη δομή της βοήθειας. Είναι αποτελεσματική όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, τα χρήματα των φορολογουμένων αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο. Στι συζητήσει μας σήμερα θα εξετάσουμε διάφορες εναλλακτικέ και μοντέλα. Θα εξετάσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η βοήθεια να μπορεί να λειτουργεί όπως πρέπει και να εξετάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες τα φτωχά κράτη κατάφεραν να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Έχουμε εδώ έναν εμπειρογνώμονα, τον κύριο Ρούντι Ντελαρού από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Θα έρθει σε πέντε λεπτά. Έχουμε όμως και, τον, και την εισηγήτριά μας, την κυρία Θεοχάρους, και θα της δώσω το λόγο, ενώ περιμένουμε να έρθει και ο κύριος Ντελαρού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω το λόγο. You have the, Έχετε το λόγο, ναι. Να ξεκινήσω με ένα μύθο της πατρίδας μου. Ένα μύθο από την αρχαία Ελλάδα. Είναι ο μύθος των Δαναίδων. Οι Δαναίδες ήσαν οι 50 κόρες του βασιλιά Αίγυπτου που έδωσε και το όνομά του στην Αίγυπτο. Αυτός πάντρεψε τις 50 του κόρες με 50 πρίγκιπες παρά τη θέλησή τους και αυτές συμφώνησαν ένα βράδυ και τους σκότωσαν όλους και η τιμωρία από τους θεούς ήταν να προσπαθούν να γεμίσουν ένα πίθο ο οποίος είχε χιλιάδες τρύπες επάνω με νερό και κουβαλούσαν με τα κανάτια και κουβαλούσαν για να γεμίσουν αυτό τον πίθο. Η Αφρική και ο αναπτυσσόμενος κόσμος είναι ο πίθος των Δαναίδων με χιλιάδες τρύπες που προσπαθούμε να τον γεμίσουμε με νερό χωρίς να έχουμε κλείσει πρώτα τις τρύπε. Και βεβαίως οι 50 Δαναίδες μπορεί να είναι σήμερα και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσω, θα συνεχίσω λέγοντας σας ότι η οποιαδήποτε βοήθεια προς τους λαούς που θα παρασχεθεί θα πρέπει να δίδεται με απόλυτο σεβασμό και λαμβάνοντα υπόψη ότι υπάρχει τρομερή καχυποψία ανάμεσα σε αυτού του λαού εναντίον των Ευρωπαίων γιατί του θεωρούν υπεύθυνου για πολλά από τα δεινά τα οποία έχουν υποστεί αλλά και μια επακτωμένη νοοτροπία να θεωρούν επίση ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη να του συντηρήσει, είναι υπεύθυνη να του ταΐσει, είναι υπεύθυνη να του βοηθήσει στην ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι απόλυτο και δεν ισχύει για όλου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει, ένα γενικό, έχει μια γενικότερη ας πούμε, εφαρμογή. Το τρίτο θέμα είναι τα διαθέσιμα ποσά. Γνωρίζουμε κάθε χρόνο ποιο είναι ο προπολογισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι ο προπολογισμό για την, το, το eradication of poverty, το alleviation of poverty από, τις, από τα κράτη-μέλη. Ε, σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να λάβουν μέρος βέβαια και η κοινωνία των πολιτών με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Χτες έμεινα έκπληκτη ακούγοντας την σχέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις γιατί νόμιζα ότι αυτά τα θέματα είναι ξεκαθαρισμένα εδώ και καιρό. Αν πρέπει να ρυθμίσουμε το Συμβούλιο, την διοίκηση, τον προπολογισμό, του στόχου μια NGO, μια μη κυβερνητική οργάνωση, τότε πάβει να είναι μη κυβερνητική οργάνωση και αν του δίνουμε περισσότερα λεφτά από ένα συγκεκριμένο ποσοστό του προπολογισμού του, του μετατρέπουμε σε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό τέρα, το οποίο σίγουρα θα απασχολεί πολλού, αλλά δεν θα προάγει εκείνο που είναι ο στόχο του, την κοινωνία των πολιτών και την εθελοντική δράση. Γι' αυτό πραγματικά χτε δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά, συγχωρέστε μου την άγρια, αλλά νομίζω ότι ήταν τρομακτικά έξω από την γραμμή αυτά που λέγονταν όσον αφορά τις NGO. Ναι, οι NGO έχουν ένα τρομακτικό ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η φτώχεια δημιουργεί φαύλους κύκλους, μέσα στους οποίους εμπλέκεται η νόσηση, κυρίως η, ε, ε, η νόση που μεταδίδονται με ε, σεξουαλικά, όπως είναι το AIDS και άλλες sexually transmitted diseases, είναι η μετανάστευση, η μη ελεγχόμενη μετανάστευση, η δημιουργία κακών συνθήκων παροχής ε, ε, υπηρεσιών υγείας, η εγκληματικότητα και όλα τα συναφή. Άρα εμείς πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο αυτό σε κάθε περίπτωση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια. Για παράδειγμα, το AIDS ξεκίνησε ως μια νόσος περιθωριακών ανθρώπων, τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι η νόσος των φτωχών. Άρα πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο εκεί ακριβώς που είναι και ο πιο αδύνατος. Για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι είναι το κυριότερο και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που να έχουν σχέση οπωσδήποτε με την ε, δημιουργία ενεργειακών πηγών, ανανεωσίμων επιτοπλίστων, υπηρεσιών υγείας, όσον αφορά την, τα σχολεία και την εκπαίδευση, όσον αφορά την παροχή ποσίμου νερού και όσον αφορά την διαχείριση των λιμάτων και των αποχετεύσεων. Βεβαίω, βασική προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση και η παραμονή των ε, επαγγελματιών στη χώρα τους και η μη απομίζηση τους προς την Ευρώπη και την Αμερική. Είναι η εκπαίδευση στην δημοκρατία, είναι η εκπαίδευση στη σωστή διακυβέρνηση και είναι και οι ειδικέ ηθίκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Αυτά ως ένα γενικό περίγραμμα, βεβαίως μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Τίθεται και ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι, αν η βοήθεια θα πρέπει να δίδεται αδιακρίτως και σε χώρες οι οποίες ενώ έχουν τεράστια ε, ποσοστό του πληθυσμού τους ζει στην απόλυτη φτώχεια, καταγίνονται με το πώς να φτιάξουν πυρηνικά όπλα, δαπανούν τεράστια ποσά στο να φτιάχνουν πυρηνικά όπλα ή να αποδίδονται σε εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς. Εκεί είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα σταθμίσουμε και την προσέγγιση μας. Βασικά πιστεύω ότι όλα όσα έχουμε πει και έχουμε μάθει μέχρι σήμερα είναι σημαντικά και πάνω σε αυτή την εμπειρία θα οικοδομήσουμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για να αποφύγουμε την διαφθορά, την κυβερνητική, την έλλειψη δημοκρατία θα πρέπει να εστιάσουμε στην κοινότητα, στι μικρέ κυψέλε ανάπτυξη, οι οποίε θα βοηθήσουν εκ των κάτω προ τα πάνω να αναπτυχθεί και η δημοκρατία και τα δημοκρατικά Ινστιτούτα και η σωστή διακυβέρνηση, αλλά πρωτίστω οι καλύτερε υπηρεσίε προ τον λαό, οι καλύτερε υπηρεσίε προ του ανθρώπου. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κατά μέγιστο 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε αργήσει. Thank you for uh, the invitation. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Πρόεδρος, κύριε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Εκ μέρους του κυρίου Σομαδία, ε, του Διευθυντή, την Επιτροπή Ανάπτυξης που με κάλεσε. Εμείς της ε, ΔΟΕ είμαστε μια τριμερής οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών και έχουμε μια εντολή που είναι πολιτική, ρυθμιστική και τεχνική ταυτόχρονα. Και η αναπτυξιακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για την πρόθεση της ε, αξιοπρεπούς εργασίας. Σε αυτό θα επανέλθω. Η Επιτροπή Ανάπτυξης το 2007 υποστήριξε το ψήφισμα για την αξιοπρεπή εργασία το 2007 και το 2006 υποστηρίξατε ένα ψήφισμα για την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης. Επίσης υποστηρίξατε και πιο ε, συγκεκριμένα θέματα ε, για την παιδική, ε, παράδειγμα για την παιδική εργασία, για την εργασία των ανηλίκων. Τώρα αυτή τη φορά είναι μια, πρόκειται για μια πρεμιέρα, γιατί το θέμα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και καλύπτει και άλλες πολιτικές διαστάσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια ενωτική αντιμετώπιση του θέματος. Θέλω να αναφερθώ στη χθεσινή συνεδρίαση της, ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Κωνσταντινούπολη, όπου ε, παρενέβη και η ΔΟΕ για τα θέματα αυτά της ανάπτυξης. Εγώ Έχω εδώ ένα αναλυτικότερο κείμενο το οποίο θα σας δώσω. Το κείμενο είναι στα αγγλικά, η περίληψή του είναι στα γαλλικά. Έχω επίσης και άλλη τεκμηρίωση στη διάθεσή μου. Και θα ξεκινήσω τώρα την τοποθέτησή μου με ένα PowerPoint. 12-13 λεπτά θα μιλήσω. Θέλω να σας ε, μιλήσω για το, διεθνές, ε, για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Απασχόληση, για την Αφρικανική κρίση ε, συνεισέφεραν και οι Αφρικανοί και να σας πω πώς μπορεί να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Διεθνές Σύμφωνο είναι κάτι που θα ήθελα να τονίσω πως ε, έχει εγκριθεί από, ε, με, με γενική συνένεση από 83 ε, χώρες. υπάρχει απόλυτη συνένεση ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Χάρη στην ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συντονισμού στο πλαίσιο του ILO Υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία παράλληλα με τις αναπτυσσόμενες χώρες και διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει σημαντικό input όπου πολλοί αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων ε, έχουν συμμετάσχει και με περιφερειακή συμμετοχή όχι μόνο της Αφρικής αλλά και της Λατινικής Αμερικής, Ασίας και Ευρώπης. Μπορέσαμε επίσης να οικονομήσουμε συνένεση στον ε, διευθυντικό όργανο το οποίο το ενέκρινε τον Νοέμβριο. Αυτοί οι τελευταίες γραμμές έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, στο πακέτο αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτή η ε, σύμβαση είναι Διεθνώ συμπεφωνημένα μέτρα πολιτικής τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο επίσης ε, αφορούν και ένα σύστημα μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη διαφορετικές καταστάσεις και σχέσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ένα βασικό ε, στοιχείο είναι ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε την, ε, τη χρονική περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στην κρίση και την ανάκαμψη. Αυτό το σύμφωνο αποτελεί την ε, απάντηση στην κρίση. Αναφέρονται 25 δυνατότητες πολίτης επιλογής σε τέσσερις τομείς που άπτονται την, της ε, απασχόλησης, του συστήματος κοινωνικής προστασίας, ε, ενίσχυσης ε, των διεθνών εργατικών προτύπων και την δήλωση τα για την κοινωνική ευθύνη, η ισότητα των φύλων και μη διακρίσεις είναι ζήτημα βασικό που καλύπτεται όμως και από τα διεθνή εργατικά πρότυπα. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα πριν από την κρίση είχαμε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και θα πρέπει να θέσουμε την απασχόληση και την κοινωνική πρόνοια στο επίκεντρο. Ως ILO έχουμε κάνει ανάλυση για, τα G, τους G20 και από τις χώρες που εξετάστηκαν οι περισσότερες έχουν προωθήσει πακέτα ανάκαμψης. Αλλά η φορολογική παρέμβαση είναι πολύ περιορισμένη στις περισσότερες από τις χώρες. σε αυτό το στάδιο πολλά κράτη χρησιμοποιούν το σύμφωνο. Έχουμε περιφερειακές πρωτοβουλίες όπως στις νήσους του Ειρηνικού. Όλες οι χώρες του Ειρηνικού έχουν παρόμοια προγράμματα και προσπαθούν να φορούσουν μια γενικότερη στρατηγική. Η Αφρική επίσης συζητάει το θέμα της περιφερειακής στρατηγικής αλλά και άλλες περιοχές. Είναι λοιπόν πολύ καλό που κράτη και περιφέρειες προσπαθούν να εξεύρουν κάποιες πιο βιώσιμες προσεγγίσεις ε, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Το ΑΕΛΟ θέλει να υπογραμμίσει πως έχουμε κάνει μελέτες ε, φυκτότητας για τα συστήματα κοινωνικής ε, πρόνοιας αυτό είναι δυνατόν να συμβεί και για τις ε, χώρες χαμηλού εισοδήματος. Χρειάζεται όμως ε, μια αλλαγή των φορολογικών συστημάτων. Επίσης, βλέπουμε ότι πολλές χώρες ε, έχουν προγράμματα για αξιοπλήρη απασχόληση. Έχουμε κάνει όμως ανάλυση ότι από τις 48 χώρες, 48 προγράμματα μάλλον που ε, αναπτύσσονται στην Αφρική, υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικών μέσων και εργαλείων. Δεν υπάρχει σύνδεση με την μακροοικονομική πολιτική χρειάζεται να στοχεύσουμε σε προσεγγίσεις ε, που αφορούν στην ανάπτυξη της εργασίας και υπάρχουν ε, και κάποια προβλήματα που δημιουργούνται από bottlenecks ε, συμφορήσεις που αφορούν τις δεξιότητες, τις ικανότητες Είναι πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να αναπτυχθεί μια στρατηγική απασχόληση χωρίς ε, την κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία αποτελεί επένδυση. Είναι ένα θέμα παραγωγικό. Και τέλος, αυτή οι αναλύσεις μας θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, να δείξουμε τις ε, ικανότητες ε, των κοινωνικών εταίρων. Θα είμαι σύντομος στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε κάνει μια νέα δημοσίευση σχετικά με τους δείκτες. Μιλάμε για δείκτες ε, αξιοπρεπούς εργασίας, αυτοί που αναφέρονται στην οθόνη είναι οι δείκτες της χιλιετίας τέσσερις δείκτες που είναι γνωστοί από το 2008. Προσπαθούμε να τους ε, εφαρμόσουν. Οι δείκτες όπως ε, το ποσοστό αύξησης ε, του εργατικού δυναμικού, η απασχόληση ατόμων που ζουν κάτω από το κατώτατο όριο διαβίωσης, Φυσικά θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αλλά μα δίνουν καλές προφορίε για την αγορά εργασία. Δουλεύουμε επίση και σε μια σειρά άλλων, με μια σειρά άλλων δικτών, θέματα σχέσεων μεταξύ εργοδοσία και εργαζομένων. Επίσης, <clears throat> και αυτό είναι ένα ζήτημα κλειδί για μας, βοηθάμε αναψώμενες χώρες με την αξιολόγηση. Έχουμε δημοσίευσαμε μία μεθοδολογία την πέντε εβδομάδα που θέλει να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κρίσης ε, στην οικονομία τους αλλά και στους μέρους κλάδους προκειμένου να γνωρίζουν πού υπάρχουν ε, ευκαιρίες απασχόλησης. Υπάρχουν επίσης και αξιολογήσεις ε, για θέματα κοινωνικής προστασίας. Μερικά ακόμα παραδείγματα. Η ανάλυση που κάναμε για το, η ανάλυση που κάναμε για το G20 δείχνει ότι οι επενδύσει στι υποδομέ είναι αποτελεσματικέ για την προαγωγή της απασχόλησης, αλλά θα πρέπει να είναι εντάσσεω εργασίας και φιλική προς το περιβάλλον. Το να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις ε, όπως ε, διευκολύσεις ε, στις πιστώσεις κλπ Πρέπει να στοχεύσουμε σε προγράμματα για τους νέους. Προσόντα. Υπάρχουν παρόμοιες παρόμοιες επενδύσεις για την εκπαίδευση στην ε, Αφρική αλλά και στην Ασία και ένα τελευταία στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω προτού να φτάσω στην Αφρική είναι το πρασίνισμα της οικονομίας είμαστε πεπισμένοι πως ε, υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες απασχόλησης πλαίσιο της πράσινης οικονομίας σε ανεψόμενες χώρες. Έχουμε προωθήσει ένα πρόγραμμα, 10, χρόνια, 10 χώρες που έχουν υπογράψει συμπεριλαμβάνουμε και λιγότερο επιτυγμένε χώρες όπως η Αϊτή, Φιλιππίνες, Σομαλία, Τανζανία και οι αναδυόμενες οικονομίες. Έχουμε παραδείγματα αναδάσωσης στην Αϊτή για την κρίση στην Αφρική έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι διαθέσιμο. Θα συζητηθεί περαιτέρω στο Ουαγκαντούγκου το Δεκέμβριο. Να αναφέρω πως ε, υπάρχει αυξανόμενη συνένεση στην Αφρική πως η απασχόληση και η κοινωνική πρόνοια είναι θέματα πολύ σημαντικά για αυτές και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στην Αφρική που να μην είναι κάτι που υπάρχει πανταχού, ότι η συνεταιρισμοί έχουν ε, μεγάλη δυνατότητα, μεγάλη δύναμη. Έχουμε επίση το θέμα των δυνατοτήτων των κυβερνήσεων και των κοινωνικών εταίρων. Γίνονται λοιπόν, υπάρχει μια συνεργασία σε διάφορα επίπεδα. προσπαθούν να υποφερθούν από τα συγκριτικά, ε, συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αφρικής αλλά παράλληλα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μεταναστευτικές ροές ε, τόσο εντός ε, Αφρικής όσο και εκτός. Τέλος, γνωρίζετε καλύτερα από μας πως ε, να συμβάλλεται αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό πως όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προάγουν την αξιοπρεπή εργασία αλλά αυτά, αυτό δυστυχώ ε, δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα, σε όλα τα έγγραφα, σε όλα τα κείμενα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταλαβαίνετε πολλά πρέπει να γίνουν. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων είναι κάτι επίγουσα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως ε, θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, την αξιοπρεπή εργασία σε διάφορους ε, τομείς όπως υποδομές, πράσινη ανάπτυξη, υγεία η υγεία θα πρέπει να συνδέεται με την κοινωνική προστασία, εμπόριο, διακυβέρνηση και αλλαγή κλίματος. Όλα αυτά λοιπόν έχουν γραφτεί σε έγγραφο της Κομισιόν του 2007 για την απασχόληση και χρειάζεται επίσης και υποστήριξη της οικοδόμησης δυνατοτήτων από τους κοινωνικούς εταίρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζήμερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλά τεκμηριωμένη παρουσίαση το του προγράμματος, του Παγκοσμίου Προγράμματος Θέσεων Εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό εμείς ως Επιτροπή Απασχόληση απασχόλησης να ασχοληθούμε εντατικότερα με το θέμα από ό,τι κάναμε κατά το παρελθόν. Έχω μία σειρά προτάσεων που πρέπει να συζητηθούν. Τίθεται πρωτίστως το ερώτημα της σύνδεσης με το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως αφού εξετάσουμε και την αποτελεσματικότητα της Συμφωνίας Κοτονού. Είπατε για παράδειγμα ότι η κοινωνική προστασία είναι από τις σημαντικότερες επενδύσεις στο μέλλον. Προγράμματα θέσεων εργασίας ε, χωρίς κοινωνική, προστασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα οι επενδύσεις, η υποδομή θα συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία απασχόλησης θέσεων εργασίας. Ξέρουμε ότι στη Συμφωνία Κοτονού, για παράδειγμα όμως, η στήριξη των επενδύσεων σε δημόσιες υπόδομες, στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών, αποκλείεται. Δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις εκεί. Το πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού δεν είναι λοιπόν το ενδεδειγμένο, υπ' αυτή την έννοια, για να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επίσης, στη συζήτησή μας κατά την ε, εξέταση της Συμφωνίας Κοτονού θα πρέπει να το δούμε αυτό ε, πολύ περισσότερο. Και έχω κάποιες προτάσεις για το πώς θα συμβάλλουμε ούτω ώστε να υπάρξει αποτελεσματική υποστήριξη για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφόρα ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τρίτον, τα ελείποντα μέσα για την εξασφάλιση της εργασίας, της κοινωνικής προστασίας αλλά και του εργατικού δικαίου έμαθα για την Παραγουάη πρόσφατα ότι ναι μεν υπάρχει καλό εργατικό δίκαιο και καλό σύστημα κοινωνικής προστασίας, αλλά η εφαρμογή του χωλαίνει σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει η νομοθεσία χωρίς να εφαρμόζεται, χωρίς να περνάει στην κοινωνική πρακτική. Εκεί χρειάζεται συγκεκριμένη βοήθεια και υποστήριξη και από έξω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση που μόλις ακούσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα και μετά από πρόσκληση σε αυτή την Επιτροπή, εγώ πήγα στο Παρίσι σε μία συνάντηση του για την απασχόληση και τη διαχείριση της κρίσης. Και ο διευθυντής ε, της ΔΟΕ, ο κύριος Σωμαδία, έθεσε το θέμα ότι η οικονομική κρίση εκφράστηκε με τη μεγαλύτερη στιγνότητα και σκληρότητα και καταστροφικά για την απασχόληση. αλλά πολλές από τις στρατηγικές για την έξοδο της κρίσης προδιαγράφονται ως στρατηγικές μείωσης της απασχόλησης. Και ο κύριος Σομαδία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εντατικής δημιουργίας θέσεων αποσχόλησης στους κλάδους εκείνους που σχετίζονται με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Εμείς δεν θέλουμε η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου να γίνει εις βάρος της απασχόλησης. Το αντίθετο θέλουμε και θέλω να ρωτήσω εμείς θεωρούμε πολλές φορές ότι στις μη αναπτυγμένες χώρες το θέμα της απασχόλησης δεν είναι πια και τόσο σημαντικό, διότι έχουμε την επίσημη και την άτυπη εργασία. Αλλά ένα από τα συμπεράσματα της συνεδρίασης στο Παρίσι, και φαντάζομαι και της ΔΟΕ, είναι το εξή ότι η κρίση έπληξε τόσο την άτυπη όσο και την επίσημη εργασία. Οπότε εμείς δεν πρέπει να βρίσκουμε άλοθη για τις αναπτυσσόμενες χώρες λέγοντας ότι έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς απασχόλησης από ό,τι οι αναπτυγμένες χώρες. Η κρίση πλήττει όλους τους τομείς. Ευχαριστώ κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, γιατί είναι η μητρική γλώσσα του προσκεκλημένου μας από το ILO. Όλο αυτό το πρόγραμμα για ανθρώπινη και αξιοπρεπή εργασία του ILO είναι πολύ σημαντικό για αυτούς που έχουν την ατυχία να ζουν σε φτωχές χώρας. Αν και υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και στις αναπτυγμένες χώρες για τους εργαζομένους. Μπορείτε να διευκρινίσετε γιατί ειδικά τώρα στην εποχή της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης η, ε, τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν μια διέξοδο από την κρίση Τώρα υπάρχουν δυνατές φωνές που ζητούν έξοδο από την κρίση. Πολλοί λένε ότι η οικονομία λειτουργεί καλύτερα όσο λιγότεροι κανόνες υπάρχουν. Από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει καλή ε, προστασία της υγείας, ε, συντάξεις αξιοπρεπής, εν πάση περιπτώσει μια σταθερότητα για το μέλλον που θα αυξάνει και την κατανάλωση. Και η υγιείς καταναλωτές είναι καλή για την οικονομία. Η κοινωνική προστασία και η ανθρώπινη αξιοπρεπής εργασία, η κοινωνική προστασία είναι λοιπόν ένα μέσον και μία διέξοδος από την κρίση. Τίθεται βέβαια το ερώτημα, ισχύει αυτό και πώς ισχύει για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ το πιστεύω. Εσείς τι λέτε. Θα ακούσουμε και λίγες ε, ακόμη ερωτήσεις. Η κυρία Ντε Κέιζερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία μου για την παρουσίασή σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δεν μπορέσατε να είστε τόσο αναλυτικός όσο θέλατε. Εγώ λοιπόν ξεφυλίζοντας το κείμενο έψαξα να βρω ποια είναι η θέση του κοινωνικού διαλόγου στην όλη διάρθρωσή σας. Διότι ένα οποιοδήποτε σύμφωνο ή μία νομοθεσία άμα δεν έχει και μία αντιστάθμιση ε, εξουσίας, ένα συνδικάτο ή οτιδήποτε, ε, ε, είναι έρμεο προστασίας. Λοιπόν, θα κάνω μία ανόητη ίσως ερώτηση, αλλά ποια είναι η διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Αφρική μπορούν να είναι ένα σοβαρό συνομιλητή στον κοινωνικό διάλογο ή είναι οι ανθρωπιστικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις που υποκαθίστανται σε αυτές τις τόσο αδύναμες ή ανύπαρκτες ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κύριος Κέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της ΔΟΕ. Οι αρχές τις οποίες αναφέρεστε είναι υπεράνω πάσης υποψίας, αλλά χρειάζεται όμως ε, και ε, λίγος βούρδουλας για να εφαρμοστούν όλες αυτές οι αρχές. Ας πάρουμε εμείς την πολινική Συμφωνία ε, τη σεβάστηκε ελάχιστα η Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη ήταν από καιρό ε, ενημερωμένες ε, για την εφαρμογή των νέων όρων αλλά στο Μπαγκλαντές χρειάστηκε να αυξήσουμε κατά 72 ώρες την διάρκεια της εργασίας για να, μπορέσουμε, να, να μπορέσει τον Παγκλαντές να αντέξει τον ανταγωνισμό. Ε, λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι ντογκελάς, λέει ο, ο μιλητής, επιτρέψτε μου την έκφραση, δηλαδή είναι έσχος στα ελληνικά. Ε, ε, όλα αυτά λύθηκαν με διαπραγματεύσεις, τα οποία κράτησε, οι οποίες κράτησαν 10 λεπτά. Θέλω λοιπόν να ξέρω πώς το περνάει το μήνυμα η ΔΟΕ. Πραγματικά δηλαδή χρειάζεται ε, ε, ένας πραγματικός καυγάς, ε, χρειάζεται μία πίεση, διότι η κατάσταση είναι κατεπίγουσα και πρέπει να αλλάξει. Επίσης, πολύ σωστά είπατε ότι η περίοδος ανάρρωσης των οικονομιών μετά την κρίση είναι 5-6 χρόνια. Αν η ανάπτυξη ξεπεράσει το 3% στις περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να αφαιρέσουμε ένα 3% για να φτάσουν, βρούμε το πραγματικό αναπτυξιακό κατόφλι, γιατί η δημογραφική αύξηση ε, ροκανίζει το, το αναπτυξιακό ποσοστό. Εσείς, στις διάφορες ρυθμίσεις σας, έχετε και μία πρακτική η οποία ονομάζεται πρόθεση των έργων με μεγάλο αριθμό απασχολωμένων. Στο Παρίσι ελήφθησαν συμφωνίες και θα υπάρξουν χώρες τις, μεγάλε μεγάλες εταιρείες της Δύσης ε, που θα αναλάβουν έργα. Ε, η ΔΟΕ είναι έτοιμη να προτείνει την ε, πρόσληψη περισσότερου προσωπικού ε, για την εκτέλεση έργων στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχετε κάνει κάποια αξιολόγηση όλων αυτών των πραγμάτων. Και τελευταίο, θέλω να επιμείνω, υπάρχει ανάγκη στις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό σύστημα. Αν ε, δεν έγινε χαμός εδώ ε, στο βορρά, γιατί δεν έγινε, διότι υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω ότι στην Αμίμπια έγινε ένα πείραμα για την ε, λειτουργία καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να ξέρω πώς λειτουργήσε το πείραμα στην Αμίμπια τι συμπεράσματα έχετε. Η κυρία Τόια έχει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη μελέτη. Και εύχομαι όλα αυτά, όλες αυτές οι ωραίες ε, γραμμές ε, και θέσεις του συμφώνου να εφαρμοστούν με τα κατάλληλα μέσα. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτο θέλω να τονίσω την ε, κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Είναι μία από τις πολιτικές που αναφέρουμε μαζί με το χρονοδιάγραμμα και άλλα. Ε, πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε πολύ πιο έντονα τις διεθνείς ε, συμφωνίες και τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ελπίζω να μην είμαι θεροβάμων, αλλά πιστεύω ότι μέσα από την ανάληψη κοινωνικής ευθύνη επιχείρησης μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ένα δεύτερο σημείο είναι ένα στοιχείο που διαφάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε μία από τις ομάδες εργασίας της ΑΚΕ και αυτό μετά από την παρουσίαση μίας μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με την τωρινή κρίση, την ε, ε, φτώχεια, την ε, πείνα και την ανεργία στις αναπτυσσόμενες χώρες και την παρουσία της ΟΗΜ που μας παρουσίασε επίσης μία μελέτη. Θέλω να ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να τα συνδέσουμε με το σύμφωνο που εσείς μας παρουσιάσατε. Εμείς ε, σήμερα διαπιστώνουμε ότι πολλοί μετανάστες ε, γυρίζουν πίσω στις χώρες τους και τελικά γυρίζουν πίσω και είναι πιο φτωχοί από όταν ε, έφυγαν διότι είχαν επενδύσει όλες τους τις οικονομίες για να φύγουν στην Ευρώπη και όταν απελάβνονται γυρίζουν πίσω είτε γυρίζουν πίσω γιατί δεν έχει πια δουλειά εδώ πέρα. Σε αυτή λοιπόν τη συνεδρίαση είπαμε ότι θα έπρεπε να μελετηθούν προγράμματα που θα πρέπει να συνοδεύονται φυσικά και από σχέδια των κρατών μελών, αλλά που θα έπρεπε να τα εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα συνοδευτικά με επιμόρφωση να δημιουργηθούν εκεί θέσεις εργασίας γιατί έστω και σε ελάχιστο βαθμό αυτοί οι μετανάστες έχουν αποκτήσει μια κάποια επαγγελματική εμπειρία που μπορούν να αξιοποιήσουν στη χώρα τους. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν και στα πλαίσια αυτού του συμφώνου ε, κάτι που να πηγαίνει σε αυτήν την κατηγορία του πληθυσμού, ο κύριος Μίτσελ. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Ντελαρού για την ε, παρουσίαση αυτή για την ε, ανεργία μίλησε, την υποαπασχόληση δεν μίλησε και πώς μετριέται. Μίλησα με έναν Υπουργό Οικονομικών Αναπτυσσόμενης χώρας που μου είπε ότι έχει πολύ υποαπασχόληση. Πώς την μετράτε την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεύτερο, ένα συνάδελφο είπε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι καλές θέσεις εργασίας με κοινωνική προστασία κλπ. Η ILO έχει εξετάσει παραδείγματα συνεταιριστικού κινήματος σε άλλες χώρες όταν πέρασαν από τη φάση της ανάπτυξης. Και επίσης ο Πατ Ντεκόπ Κάλαχερ, λέγεται Ντεκόπ, ε, ένας ευρωβουλευτής εδώ ήταν, ε, πήρε το παρονίμιο αυτό επειδή ο πατέρας του ήταν μεγάλος συνδικαλιστής. Ε, και συνέβαλε κάποια στιγμή στην ε, δημιουργία και την εδραίωση του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μου. Και τέλος, κάποια στιγμή του χρόνου, στην Επιτροπή μας θα ξαναδούμε το θέμα της ιδιοκτησίας γης και πώς μπορεί να δημιουργήσει κεφάλαιο και πώς το κεφάλαιο μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η ILO το εξέτασε αυτό το θέμα και πώς μπορεί να συμβάλλει στο θέμα που μας απασχολεί. ο κύριος Δελαρίου για να απαντήσει συνολικά σε όλες τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, ερωτήσεις ε, που ήταν ε, ε ποικίλε. Σχετικά με την εφαρμογή στην Παραγουάη, παραδείγματος χάρη, <clears throat> έχουμε ένα πρόγραμμα για την εκρίζωση της ε, παιδικής εργασίας. Το θέμα της διαχείρισης της εργασίας παραμελήθηκε σε πολλές χώρες. Η συνέπεια είναι ότι ε, ολόκληροι τομείς συρρυκνώθηκαν όχι μόνο γιατί δεν υπήρχε διοίκηση εργασίας, αλλά ε, οι αρχές ε, δεν ρύθμισαν πολλούς τομεί της αγοράς εργασίας. Είναι και αυτό ένας λόγος, ένα στοιχείο. Είναι σημαντική η εφαρμογή όλων αυτών των νομοθετικών μέτρων για την ΑΕΛΟ, γιατί υπάρχουν πολλές συμβάσεις. Όταν επικυρωθούν υπάρχει και σύστημα ελέγχου της εφαρμογής και μέσα σε ορίζοντα 5-10 χρόνια έχουμε αποτελέσματα. Αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να υπάρξουν μόνο όταν υπάρχει πολιτική δέσμευση κάθε χώρα υπέρ τη συνεργασία. Αν υπάρχει δέσμευση αυτή σε πολιτικό επίπεδο, τότε η τεχνική συνεργασία κάνει πολλά. Αν δεν υπάρχει, όπως στην Βυρμανία, όταν δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση, τότε είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, ασκούν πιέσεις, είπα κι άλλοι, καμιά φορά οι πιεσει ωφελούν, όπως στη Λευκορωσία που είναι άλλη κατηγορία χώρα, αλλά ε, εδώ υπάρχει ένα άνοιγμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Δεν είναι ο παράδεισος, αλλά υπάρχει ένα άνοιγμα. Το δεύτερο στοιχείο, ε, επίσημη, ε, ανεπίσημη απασχόληση, αυτό το έθιξαν πολύ μάλιστα, πάντοτε δουλεύαμε πάνω στη βάση της εργασίας ε, και των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τον την επίσημη ή ανεπίσημη οικονομία. Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε συστήματα μετρήσεων για να μετράμε την απασχόληση συμπεριλαμβάνοντας την άτυπη οικονομία. Το θέμα της υποαπασχόλησης είναι κλειδί σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε πάνω από 75% απασχόληση του πληθυσμού για τον απλό λόγο ότι όλοι υποχρεούνται να εργάζονται. Γιατί είναι πολύ χαμηλή μισθή και δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Ε, Όσοι οι περισσότεροι δουλεύουν κάτω από το όριο της φτώχειας, μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ορισμένο, αλλά υπάρχει και το 1,25 δολάρια τη μέρα που είναι από την Παγκόσμια Τράπεζα. Τώρα καινούριο είναι αυτό, πριν ήταν ένα δολάριο ε, σε καθημερινή βάση λοιπόν από αμοιβέ. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση στι αναπτυσσόμενε χώρε. Αν συγκρίνουμε τι βιομηχανικέ χώρε όπω τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι αναπτυσσόμενε, συνήθω διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απασχόληση είναι εκεί πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό. Αλλά είναι πολύ ευάλωτη παρόλα αυτά. Και με μία εξαίρεση το ποσοστό απασχόληση των γυναικών που είναι χαμηλό. Αλλά οι άντρε ε, δουλεύουν, απασχολούνται πολύ στι αναπτυσσόμενε χώρε. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα σε εποχές κρίσεων και γιατί θα πρέπει να αποφύγουμε τη μείωση της κοινωνικής και εργατικής προστασίας γενικότερα και της κοινωνικής. Ε, ένα τριμεμερές σώμα του ILO συνεδρίασε για πρώτη φορά στην αρχή της κρίσης και τότε εξέδωσε έξι κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα ανάκαμψης. Και το πρώτο ήταν ότι θα πρέπει να μην μειώσουμε το επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα διεθνή πρότυπα και πρότυπα εργασίας. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, τότε θα ε, καταποντιστούμε και κανείς δεν θα ανακάμψει. Μόνο θα είμαστε ε, σε ωφέλη για όλους όταν όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν την κοινωνική προστασία και την απασχόληση για όλους. Αλλιώς ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε σε φάση ανάκαμψης και όλοι θα υποφέρουν, περισσότερο δε από όλους οι φτωχότερες χώρες. Για τον κοινωνικό διάλογο. Στην Αφρική Βέβαια είναι μεικτή η εικόνα, δεν είναι παντού ίδια τα πράγματα. Όμως η καλή τεχνική συνεργασία βοηθάει. Για παράδειγμα υπάρχει ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα στους εμπειρογνώμονες, είναι γνωστό τουλάχιστον, που λέγεται διάφορο, δηλαδή πρόθεση κοινωνικού διαλόγου στη γαλλόφωνη Αφρική, που ε, άρχισε πριν από 15 χρόνια, είναι δηλαδή μακρόπνο, δεν είναι διάρκειας λίγων ετών, και ήταν επιτυχές με την έννοια ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι πιο διαρθρωμένος στις περισσότερες από αυτές τις χώρες και σε τομεακό επίπεδο. Καμιά φορά ε, πιάνουν και θέματα όπως η οικιακή απασχόληση, δεν είναι μόνο δηλαδή σε υψηλό επίπεδο εργασία, αλλά σε επίπεδο βασικό και μπόρεσαν να βελτιώσουν την συμβολή τους στις πολιτικές αποφάσεις, στη λήψη τους. Πολλά μέλουν ακόμη να γίνουν βέβαια, αλλά υπάρχουν παραδείγματα ότι, που δείχνουν δηλαδή ότι η στοχευμένη ε, υποστήριξη βοηθάει όλους τους εργαζομένους. Υπάρχουν πολλά συνδικάτα και ε, ενός εργοδοτών που καλύπτουν την άτυπη οικονομία, καμιά φορά καλύπτουν και θέματα κοινωνικής προστασίας. Στην πίστη, στο συνεταιριστικό κίνημα. Δεν λέμε ότι είναι ιδεώδης η κατάσταση, αλλά υπάρχει ένα δυναμικό βελτίωσης. Αυτό που δεν είναι καλό είναι να λέμε ότι επειδή είμαστε αδύναμοι θα πρέπει να υπάρχουν άλλα ε, ε, μέσα για μας, ε, να υπάρχουν κι άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε επίπεδο διοίκησης. Αυτό είναι λάθος, γιατί αν καταπνίξουμε από την αρχή το δυναμικό ανάπτυξης ικανοτήτων, δεν θα μπορέσει να κινηθεί ε, ανωδικά ο κοινωνικός διάλογος. Για το εμπόριο. Έχετε τρία λεπτά τώρα για την ε, ΠΟΕ. Τελείωσα σχεδόν. Για τις εργασίες ε, με μεγάλη απασχόληση προσωπικού η ΔΟΕ, το γραφείο, το προεδρείο της ε, ΔΟΕ επέστησε την προσοχή στην έλλειψη συνοχής αυτών των πολιτικών. Το 2008 είχαμε μια πολιτική συμφωνία για να αλλάξουμε το καταστατικό μας και ο σύνδεσμος, ο δεσμός μεταξύ εμπορίου και εργασίας έγινε δεκτός από τις 185 χώρες. Και θέλουμε εμείς να αναλύσουμε καλύτερα την επίπτωση του εμπορίου στην εργασία και αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις. Ακόμη βρισκόμαστε στην αρχή και είναι και χρονοβόρο, χρονοβόρα όλη αυτή η διαδικασία, αλλά προσπαθούμε. Έχουμε ήδη συντάξει και ένα εγχειρίδιο σχετικά και είχαμε και μία σχετική επιτυχία. Για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων προσπαθούμε να έχουμε μία καλύτερη εφαρμογή και θέλουμε να έχουμε μία καλύτερη εφαρμογή των διαφόρων όρων ε, από τις επιθεωρήσεις εργασίας. Κοιτάστε, πρέπει να σταματήσουμε. Αυτός είναι ο χρόνος μας. Το λόγο τώρα έχει η Κομισιόν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω πως ε, συνεργαζόμαστε στενά με το ILO και πως ε, στηρίζουμε τις εργασίες τους φυσικά ειδικά την ατζέντα για την αξιοπρεπή απασχόληση και για το σύμφωνο απασχόληση. Υπάρχουν και κάποια έγγραφα γενικότερη πολιτική πάνω στο θέμα τη απασχόληση, ειδικά το συμπέρασμα του Συμβουλίου για την προαγωγή τη απασχόληση σε αναπτυσσόμενε χώρε ή για την αξιοπρεπή απασχόληση στι χώρε αυτέ. Ε, θέλαμε να πούμε ότι η Κομισιόν στι αναπτυσσόμενε χώρε προωθεί τον πολιτικό διάλογο σύμφωνα με την ατζέντα της ΆΚΑ για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας ε, και υποστηρίζει τους ε, μηχανισμούς ε, βοηθείας που είναι πλέον ευθυγραμμισμένοι με τις εθνικές πολιτικές. Εργαζόμαστε επίσης σε συνεργασία με άλλους εταίρους, ιδίω με την Διεθνή Τράπεζα. Συνεργαζόμασταν και με τον ΩΣΑ και το ΠΟΒΝΕΤ e κατά πολέμηση της ε, Ένδειας, αναφέρθηκε προ Έχει συντάξει και ένα κείμενο για την προαγωγή της απασχόλησης και την ε, κοινωνική προστασία όπου αναφέρονται φυσικά και οι επιπτώσεις ε, που υπάρχουν για τους διάφορους εταίρους. Να υπερθυμίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε και μια άμεση απάντηση στην κρίση με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επί του θέματος και την σύσταση του Vulnerability Flex με ένα συνολικό ποσό προϋποδότησης 500 εκατομμύρων ευρώ όπου ένα σημαντικό ποσό έχει δοθεί σε 17 κράτη που τους επιτρέπει να υποστηρίξουν την κοινωνική πολιτική και τους κοινωνικούς εταίρους. Να επενθυμίσω επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 2010 πρόκειται να γίνει η διάμεση αναθεώρηση του ΜΙΦΕΔ και στόχος είναι να επανεξετάσουμε με το σύνολο των χωρών του ΦΕΔ ε, τις σφαιρικές πολιτικές και ειδικά των θέση που αποδίδουν στην απασχόληση, την αξιοπρία απασχόληση και την προστασία των εργαζομένων. Να υπενθυμίσω επίσης πως μετά από τη διάσκεψη του Λισαβόνα 2007 συστάθηκε μια εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που ε, αφορά ιδιαίτερα στον τομέα της ε, κινητικότητας, της μετανάστευσης και την απασχόληση και ε, αφιερώνει μεγάλο κομμάτι στην απασχόληση. Συμπερασματικά λοιπόν να υπενθυμίσω για να επανέλθω σε αυτό που αναφέρθηκε για την αξιοπρεπή απασχόληση, σε αυτήν την έννοια της αξιοπρεπούς απασχόλησης, όπως είπε ο κ. Ντελαρή, το θέμα της ε, απασχολησιμότητας, ε, συγγνώμη όχι της απασχόλησης, θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το επίπεδο ένδυας. Ε, το ποσοστό απασχόληση είναι πιο μεγάλο στις αναψώμενες χώρες, απλά διότι ε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά για ανάμεσα στα άτομα τα οποία έχουν μια χαμηλόμιστη εργασία από αυτούς που δεν έχουν καμία. Τώρα, το, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον άτυπο τομέα της οικονομίας είναι, υποεκπροσωπούνται στον πολιτικό διάλογο και εδώ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε αυτό τον πολιτικό διάλογο και τέλος το θέμα των, ε, αρμο... των ικανοτήτων, των προσόντων, οι χώρες ε, ε, αναπτυγμένες προωθούν τη νέα οικονομία και παρατηρούμε όμως στις αναπτυσσόμενες χώρες αυτές οι νέες δεξιότητες, τα νέα προσόντα λείπουν, πρέπει να κατευθυνθεί περαιτέρω προσπάθεια στις, ε, στην εκπαιδευτική πολιτική τους για να μπορέσουν να ετοιμάσουν την μελλοντική τους ανάπτυξη επιτρέποντας σε μια γενιά να αποκτήσει προσόντα που θα τους επιτρέψει να οδηγήσουν τη χώρα σε μια καλύτερη ανάπτυξη. Ο εισηγητής μας, εισηγητή μας, συγγνώμη, κυρία έχει τον λόγο για δύο λεπτά για τα τελικά της συμπεράσματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά ενδιαφέροντα τα οποία και θα ε, συμπεριλάβουμε στο report, θα τα λάβουμε υπόψη. Βεβαίως επισημένο μία τάση να συμπεριφερόμεθα κατά κάποιον τρόπο ηγεμονικά προς τον τρίτο κόσμο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ίσως θα πρέπει να το αποφύγουμε γιατί θα δημιουργήσει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή πριν δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας προσπαθούμε να μανιπουλάρουμε τις διαδικασίες της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ. Merci. Je remercie. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη, τον εμπειρογνώμονά μας και την εισηγήτρια για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όταν η έκθεση θα ολοκληρωθεί, θα επανέλθουμε. Αναβίβολα, αυτό θα συμβεί γύρω στα τέλη του έτους. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά την αλληλεία στο Μαρόκο, σημείο 12 της Σημερισίας διατάξεως. για τη συζήτηση αυτή της νομοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας. Η συνεδρία θα διεξαχθεί και κλεισμένων το θυρών. Μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η βοηθή των μελών, η υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων που παρακολουθούν τις εργασίες της ομάδας της Επιτροπής ΔΕΔΕ και Αλίας. Παρακαλώ λοιπόν όλους τους άλλους να εγκαταλείψουν την αίθουσα και ζητώ από τους κλητήρες να διασφαλίσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της συνεδριασιός μας.